επιτευχθεί μια συνένεση όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις προς όφελος των πολιτών του Μπαχρέιν. Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε. Η συζήτηση για την κατάσταση του Μπαχρέιν ολοκληρώθηκε. Θα ψηφίσουμε μετά την εξέταση του τελευταίου θέματος στην ημερήσια διάταξη. Το θέμα αυτό αφορά την περίπτωση τη Ραφά έτσι στη Συρία. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μπιέλανη. Ευχαριστώ, Υπάρχουν διάφορες δικτατορίες στις αραβικές χώρες, αλλά σε αυτήν τη χώρα πιο συγκεκριμένα έχουμε κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ράφα Ναχέντ είναι μια ψυχαναλήτρια πολύ γνωστή στον κόσμο. Το κίνημα ελευθεριών της Συρίας έχει συνειδητοποιήσει ότι το σκηνή έχει παρατραβήξει διότι παραβιάζονται όλες οι μορφές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προσπαθούμε να το κράτος προσπαθεί πια με παρανοϊκό τρόπο να σταματήσει οποιαδήποτε κοινωνική δραστηριότητα. Δηλαδή όταν έχουμε πούμε, πειραματικά εργαστήρια συζήτησης, ε, συναντήσεις. Το ίδιο λοιπόν ε, ε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο καταστολής έπεσε και η Ράφα Νασέντ. Πρέπει λοιπόν να την βοηθήσουμε. Ο κύριος Μαστάλκα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι υπέρ της ε, απελευθέρωσης της κυρίας Ραφάνα Σέτ. Υποθέτω ότι είναι αθώα, παρόλο που μου είναι ε, δύσκολο να ε, πιστέψω τι έχει γίνει ακριβώς λόγω αυτών των παραπιστικών, παραπλανητικών εκστρατιών. Νομίζω ότι στη Συρία μπορούμε πλέον να μιλούμε για έναν εμφύλιο. Ο, η χώρα παίρνει υποστήριξη από το εξωτερικό και εμείς υποστηρίζουμε όλα αυτά τα φαινόμενα χωρίς να γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν εξεγερθεί. Η υποστήριξή μας προς την ε, Ραφά Νασέντ είναι υποστήριξη προς μια εκστρατεία υποκίνησης του μίσους. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι υπέρ της ειρήνης, άρα να καταψηφίσουμε το ψήφισμα για την κυρία Νασέτ. Ευχαριστούμε, κύριο Σταβάρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά πρώτον, ήθελα και εγώ να χαιρετήσω τους επισκέπτες ε, στο ημικύκλιο από τη Συρία που είναι στατευμένοι και υπερασπιστές της κυρίας Νασέντ. Η συζήτηση λοιπόν, λοιπόν για τα ανθρώπινα δικαιώματα δυστυχώ γίνεται τόσο αργά που δείχνει ότι δεν επιτρέπει στου συναδέλφου να παρευρίσκονται. Θα πρέπει η αίθουσα εδώ να είναι γεμάτη, γιατί μιλάμε για ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση άμεσα και πολλέ φορέ η δική μα συζήτηση οδήγησε στην απελευθέρωση κάποιων από του ανθρώπου για του οποίου μιλήσαμε παρόλο που δράση αναλαμβάνεται εκτό τη δική του τη χώρα. Ξέρουμε για τι χώρε που έχουν περάσει από δικτατορίε όπω η δική μα ότι δεν πρέπει κανεί να εγκαταλείπει του αντιφρονούντε στην τύχη του. Εδώ λοιπόν για την ε, Σύρι, Σύρια ε, ψυχαναλήτρια ε, έκανε ταξίδι προς το Παρίσι για να επισκεφτεί τη φίλη της, την κόρη της συγγνώμη, και συνελήφθη από τις αρχές της χώρας μας γράφει, και εδώ θα περάσω στα γαλλικά, ανακαλύπτω ένα κρυμμένο κομμάτι της κοινωνίας στην οποία ζω και για την οποία είμαι υπεύθυνη. Θεωρώ αξιοθαύμαστα τα λόγια αυτά τη κυρία Νασέτ. Θεωρώ ότι είναι συνυπεύθυνη για την κατάσταση στην οποία έχει φτάσει η κοινωνία τη χώρα τη. Μιλάμε για εκατοντάδε ε, ε, νεκρούς, ε, τραυματίες, ε, φυλακισμένους, πρόσφυγες στο Λίβανο, στην Τουρκία και στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια των μηνών αυτών. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει αποφασιστική δράση και να δει τι συμβαίνει με του στρατευμένου ε, του αντιφρονούντε και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία. Δεν μπορεί να έχουμε εδώ διπλά μέτρα και σταθμά. Θα πρέπει να μιλάμε με την ίδια επιμονή και την ίδια πυγμή για τα θέματα των ε, σύρων πολιτών, όπως για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Μπαχρέν και την, ε, το Θιβέτ. Η επίτροπο, ως εκπρόσωπος της ε, κυρίας Άστον, θα πρέπει εδώ να μας πει την άποψή της με σαφήνεια. Κυρία Ντεκάιζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς σήμερα το πρωί είχαμε ένα πολύ πολιτικό ψήφισμα για τη Συρία. Για τη Συρία και την Αίγυπτο και αν εμείς σήμερα το απόγευμα θελήσαμε να έχουμε ένα διαφορετικό ψήφισμα για τη Ράφα Ναζέντ, το κάναμε γιατί είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από πολιτική περίπτωση. Είναι θέμα πολιτικών δικαιωμάτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται για μια γνωστή ψυχαναλήτρια, 66 χρονών, αναρώνει από έναν καρκίνο, είναι καρδιοπαθής, είναι σε ένα κελί με άλλους 14-15 κρατούμενους σε ένα κελί και κυρίως δεν έχει κάνει και τίποτα. Πρόκειται λοιπόν ε, για αυτήν την κλασική τυπολογία πολίτη που μπορεί να είναι δημοσιογράφοι, επιστήμονες, φύλαρχοι ε, που αποδεικνύει ότι τελικά κανένας ε, δεν είναι προστατευμένος από την αυθαιρεσία. Και βέβαια εμείς ε, δεν έχουμε μεγάλες, ε, δεν έχουμε μεγάλες δυνατότητες επιρροής στη Συριανή κυβέρνηση αλλά στους φίλους της ναι ας πούμε στην Κίνα, Σαουδική Αραβία, ε, στον Αραβικό Σύνδεσμο εκεί να παρέμβουμε ούτως ώστε οι ανθρωπιστικές τουλάχιστον οργανώσεις να μπορέσουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και παρακαλώ η κυρία Ράφαν, ζητώ η κυρία Ράφα Νασέντ να απολευθερωθεί. Η κυρία Άστον επίσης έχει κάνει δηλώσεις. Μέχρι και Κάρλα Σαρκοζία έστειλε σχετική επιστολή. Λοιπόν, και εμείς ας πούμε σήμερα στη Συριακή κυβέρνηση φτάνει. Με συγχωρείτε. Πρόεδρε, Επίτροπε Κρούς, συνάδελφοι. Η κυρία Νάσεντ δείχνει το πρόσωπο των ανθρώπων που ε, στο σκοτάδι ε, πρέπει να υποστούν τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λογοκρισία στη Συρία. Βλέπουμε στο διαδίκτυο την αδικαιολόγητη και πέρμετρη κυβερνητική βία κατά των διαμαρτυρόμενων Σύρων πολιτών. Ε, όλοι όμως διακινδυνεύουν την ζωή τους προκειμένου να εκφράσουν ελεύθερα τη ζωή τους, να πούν την ιστορία τους. Αλλά μπορεί να, πυροβολ... να τους πυροβολήσει ένας ελεύθερος σκοπευτής. Παιδιά τα οποία ακροτηριάζονται, βασανίζονται και αναγκάζονται να σιωπήσουν. Παιδι... οι οποίοι παίρνουν τα πτώματα των παιδιών τους και πρέπει να τα θάψουν και να τα κρύψουν. Στην σιωπή με κηδείες οι οποίες είναι παράνομες. Οι άνθρωποι εκεί είναι σε κατάσταση θυμού και οργής που ξεπερνάει κάθε όρια. Η διεθνή κοινότητα δεν έχει συγκεκριμένη εντολή επειδή η Κίνα και η Ρωσία δεν συμφωνούν με το ψήφισμα του ΟΗΕ. Όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει και πρέπει να κάνει περισσότερα. Εδώ πρέπει να καλέσουμε έρευνα από διεθνέ ανεξάρτητο δικαστήριο για τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί. Επίση, θα πρέπει να υπάρξουν στοχευμένε κυρώσει για όσου παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είμαστε βασική εμπορική εταίρη τη Συρία. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε στοχευμένε κυρώσει για τι οικονομικέ ανάγκε τη κυβέρνηση και να του δώσουμε μια σαφή επιλογή. Ή ε, εμπορικέ σχέσει με την Ευρώπη ή απελευθέρωση με την απελευθέρωση της Ραφέντ Νασάντ ή όχι. Εδώ λοιπόν δεν μπορούμε να αφήσουμε την κατάσταση του λαού της Συρίας στα χέρια των ε, καταπιεστών. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Τουρκία για να πάψει αυτή η ανίποτη βία στη Συρία. Ναι. Ευχαριστούμε κύριο Πρέντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ επίσης θα ήθελα να απαιτήσω την άμεση απελευθέρωση της κυρίας Ραφάνα Σέιτ, πρώτης ψυχαναλήτριας στη Συρία, η οποία συνελήφθη αυθαίρετα ε, το Σεπτέμβριο και έκτοτε κρατείται παρόλο που είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση της υγείας της. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες κατηγορίες εναντίον της. Στον τύπο αναφέρεται ότι την κατηγορούν ότι είχε κάποιες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν την Συρία. Ε, και πραγματικά η κατάσταση είναι εντελώς ε, σουρεαλιστική γιατί το καθεστώς αυτό συλλαμβάνει μια ψυχαναλήτρια επειδή βοηθάει εκείνους που θέλουν να ξεπεράσουν το φόβο τους. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι η καταστολή στη Συρία δεν γνωρίζει όρια. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει αυτό το κατεπήγον ψήφισμα το οποίο συνοδεύεται από ένα κείμενο που καταδικάζουμε ξεκάθαρα αυτή την καταστολή και καλούμε τον Άσαντ να εγκαταλείψει την εξουσία του να σπάρξει μια δημοκρατική μετάβαση. Και τώρα οι ομιλητέ των πολιτικών ομάδων, η κυρία Μπασέσκου εκ μέρου του ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το καθεστώς τα καθεστώτα μάλλον που είναι δικτατορικά συχνά λαμβάνουν μέτρα κατά των ψυχολόγων και της ψυχολογίας. Εδώ καταστρέφεται η κοινωνία της Συρίας. Το 1977 αποφασίστηκε όλες οι σχολές ψυχολογίας να καταργηθούν από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και οι ειδικοί είτε καταδικάστηκαν είτε ξαναγκάστηκαν σε αναγκαστική εργασία για την κυρία Νασέτ. Λοιπόν, το καθεστώς της Συρίας συνεχίζει απλώς αυτή την παράδοση και αποδεικνύει ότι δεν είναι δημοκρατικό η Ραφανασέντ δεν είχε πολιτική δραστηριότητα, όμως η υπόλοιπη δράση της θεωρήθηκε ανατρεπτική. Και αυτά μόνο και μόνο γιατί ασχολείται με την ψυχή του ανθρώπου. Και η ψυχή έχει πάντοτε μία φυσική τάση να θρώσκει προς τα ψηλά, άνω, προς την ελευθερία. Εδώ λοιπόν Πρέπει αμέσω να αναλάβουμε δράση. Όχι μόνο γιατί η κυρία Νασιώτη ήταν μεγάλη επιστήμονα, γιατί έχει ευαίσθητη υγεία, αλλά γιατί θα πρέπει να μπορεί ελεύθερη να ασκεί το επαγγελμά τη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Σένισελ εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, η, η Ραφάνα Σάντετ συνελήφθη εντελώ αυθαίρετα το Σεπτέμβριο στη Δαμασκό, ενώ ασκούσε την ψυχανάλυση εδώ και πολλά χρόνια και βοηθώντας με τον τρόπο αυτό τα θύματα του καθεστώτος. Η πρόθεση, η, κατηγορή, η, η σύλληψη της κυρίας Νασέτ παραβιάζει κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει να ζητήσουμε άμεσα την απελευθέρωσή τη. Οι υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά του χωρί να φοβούνται κυρώσει από τι αρχέ. Σύμφωνα με τη συνθήκη τη Λισαβόνα, η υπεράσπιση των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι μια προτεραιότητα στη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις άλλες χώρες και θα πρέπει να εφαρμόζουμε σοβαρές κυρώσεις έναντι χωρών που, που παραβιάζουν κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα η κυρία Όλαντ εκ μέρους των Φιλελεύθερων και Δημοκρατών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η σύλληψη της κυρίας Νασέτη στη Δαμασκό ήταν ένα μια απόδειξη των αυθαίρετων και δύο μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση της Συρίας κατά του ίδιου του λαού. Είναι ένας από τους πολλούς που φυλακίστηκαν από τις αρχές για ισχυρισμού ε, παράνομων δράσεων που ε, δήθεν ε, σταθεροποιούν το κράτος. Εδώ λοιπόν έχουμε ψευδείς κατηγορίες οι οποίες αποδεικνύουν ότι το καθεστώ του Πρόεδρου Χαλσάν είναι κατασταλτικό για τις ελευθερίες του κάθε Σύρου πολίτη δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά μεταξύ ίκτου και αντιπαράθεσης εδώ. Εδώ η, ε, η αυξανόμενη παρανοϊκή συμπεριφορά των αρχών της Συρίας δείχνουν ότι θα πρέπει κατά τη δική τους άποψη όλες οι κυβερνήσεις να φοβούνται το λαό τους. Όμως στην πραγματικότητα το αντίθετο θα πρέπει να ισχύει. Ο λαός να μην φοβάται την κυβέρνησή του. Η κυβέρνηση της Συρίας έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ο πρόεδρος θα πρέπει να πάυσει τις πράξεις βίας και να παραδώσει την εξουσία στο λαό του έτσι ώστε να υπάρξει μια δημοκρατική μετάβαση για τη χώρα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Όγιουλαντ. Ο κύριος Καμίνσκι για τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές. E, για το θέμα της κυρίας Νασέντ είναι κάτι το οποίο ε, μας απασχολεί ιδιαίτερα εδώ στο σώμα ασχέτως από το που καθόμαστε στο ημικύκλιο όλοι πραγματικά στεναχωριόμαστε για αυτή τη γυναίκα και θέλουμε να, ελευθερωθεί. Εμείς πέρα όμως από αυτή την περίπτωση μιλάμε για τη δημοκρατία συνολικά στην Συρία. Εμείς με την αραβική άνοιξη είμαστε μάρτυρες μίας ιστορικής στιγμής. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε στεγανά και να λέμε ότι ορισμένοι ναι, έχουν δικαιώματα δημοκρατίας και άλλοι όχι και οι αδερφοί μας οι Άραβες έχουν και αυτοί δικαίωμα. Ευχαριστούμε κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση της κυρίας Ράφανα Σέντ αποτελεί σύμβολο. Η κυρία Νασέτ συνελήφθη ενώ ερχόταν στο Παρίσι για να ε, παρευρεθεί στην γέννα της κόρης της. Η κυρία Νασέντ είναι ένα σύμβολο. Είναι το σύμβολο της φοβερής καταστολής στη Συρία. Κατά όλων αυτών των ειρηνικών διαδηλωτών που όλοι είναι εντελώς αθώοι. Χιλιάδες άτομα είναι φυλακισμένα, χιλιάδες δολοφονούνται και αυτό γιατί τολμάνε να φωτογραφίζουν την καταστολή. Είναι αυτές οι, αυτές οι φωτογραφίες που εμάς μας ενημερώνουν, τις πληρώνουν με τη ζωή τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μιλάει όμως τόσο δυνατά και ανεπαρκώς ε, και, και, και ανεπαρκείς οι διαμαρτυρίες. Μόνο η πίεση στη Συριανή αστική τάξη μπορεί να ανατρέψει τον ε, Μπασέρα Σάντ. Ευχαριστούμε και τώρα ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση στη Συρία είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Ο Ασάτ παραμένει στην εξουσία λόγω της στρατιωτικής ε, δύναμης και οι επαναλαμβανόμενες ειδήσει για κατάπνιξη των διαδολιώσεων ε, αποδεικνύουν ότι οι θύνοντες ε, γίνονται όλο και πιο, έχουν όλο και πιο σπασματικές αντιδράσεις. Η αυθαίρετη σύλληψη της Νασέτ που είναι 66 ετών και είναι καρδιοπαθής και αναρώνει από καρκίνο είναι μια απόδειξη ότι οι αρχές φοβούνται και την ίδια τους τη σκιά. Ε, ε, ε δεν θα πρέπει να αναμένουμε ανθρωπισμό εκ μέρους του Συριακού καθεστώτος. Ε, η Συρία βλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν εχθρό. Ίσως μια πίεση από τη Μόσχα ή το, ή το Πεκίνο μέσω της διπλωματίας θα μπορούσε να έχει περισσότερα αποτελέσματα η υπηρεσία εξωτερική δράση θα έπρεπε να φανεί πιο επινοητική και να συνεργάζεται όχι με τους παραδοσιακούς της εταίρους. Ευχαριστούμε κύριο Έντενμπεργκ. Κυρία Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι διαμαρτυρίες στη Συρία δεν θα πρέπει να πάψουν ε, μέχρι να αντλήσουν τα διδάγματα της Αραβικής Άνοιξης οι αρχές της χώρας. Μιλάμε στην, ε, στη σημερινή, στο σημερινό θέμα για την πρώτη γυναίκα ψυχαναλήτρια της ε, χώρας που έχει βοηθήσει το λαό αυτό να ξεπεράσει τους φόβους του. Έχει οργανώσει σεμινάρια, εργαστήρια δωρεάν για τους πολίτες της χώρας και για αυτό το λόγο συνελήφθηκε στη Δαμασκό, στο αεροδρόμιο στις 10 του Σεπτέμβρη. Ακούστηκαν πολλές φωνές έκκλησης προς το καθεστώς της Συρίας ώστε να απελευθερωθεί. Και η Διεθνής Ένωση Ψυχαναλυτών ε, εξέφρασε την ίδια έκκληση, αλλά κρατείται ακόμα. Δεν ξέρουμε τίποτα για την κατάσταση της υγείας της. Η κατάσταση στη Συρία είναι απελπιστική, είναι κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει λοιπόν το καθεστώς της χώρας να συνειδητοποιήσει ότι το να ποδοπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα σημαίνει ότι θα καταδικαστεί αργά γρήγορα από την διεθνή κοινότητα. Η αλλαγή είναι αναπόφευτη και αναπόδραστη. Δεν μπορεί η βία να συνεχίζει μέρα με τη μέρα. Το είδαμε και από την περίπτωση του Καντάφη. Το τίμημα θα είναι πάρα πολύ ψηλό κάποια στιγμή. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πορέμπα. Τα πρόσφατα συμβάντα στη Συρία δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ειρηνικής επανάστασης σε αυτή τη χώρα και οι αρχές θα συνεχίσουν να αποδοπατούν και να καταστέλουν την αντιπολίτευση. Οι άνθρωποι κρατούνται ε, παράνομα. Ε, η Ραφάνα Σέντ επίσης κρατείται παράνομα. Συνελήφθη το Σεπτέμβριο στη Δαμασκό η περίπτωσή τη θα πρέπει να λυθεί άμεσα διότι και θα πρέπει ήδη να απελευθερωθεί γιατί η κατάσταση υγεία της επιδεινώνεται συνεχώς. Θα πρέπει να απευθύνουμε μία έκκληση στη Συρία να θέσει ένα τέλος αυτή την αυθαίρετη κράτηση της κυρίας Νασέτ. Επίση, να απελευθερώσει όλους τους αντιφρονούντε. και να δευκρινίσει ακριβώς να δώσει στοιχεία για την κατάσταση των ανθρώπων που κρατούνται στη χώρα αυτή. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω 18 ονόματα ε, στον κατάλογό μου για την διαδικασία Catch the Eye. Ε, θα πρέπει να επιλεγούν ε, πέντε ομιλητές. Θα ξεκινήσουμε από την κυρία Σάια. Κύριε Πρόεδρε, η Αραβική Άνοιξη είχε σαν αποτέλεσμα την ε, βία αντίδραση των Συριακών Αρχών. Μια τέτοια περίπτωση είναι η περίπτωση της κυρίας Νασέτ, η οποία συνελήφθη στις 10 Σεπτεμβρίου του 2011 ε, ε, επειδή παρήχε θεραπευτική αγωγή σε θύματα ψυχολογικών τραυμάτων. Η Συρία υφίσταται ένα δικτατορικό καθεστώς. Και ε, η κυρία Νασέτ προσπάθησε να απελύνει τις επιπτώσεις της πολιτικής αυτού του καθεστώτος. Ε, βλέπουμε στην περίπτωση αυτή και μία παραβίαση των διεθνών ε, κανόνων. Θα πρέπει αυτή η μεμονωμένη περίπτωση πραγματικά να δοθεί στη δημοσιότητα. Ο κύριος Παλέτσκης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επανειλημμένως στις συζητήσεις μας έχουμε εκφράσει την καταδίκη μας κατά του καθεστώτα της Συρίας, όμως αυτό δεν φαίνεται να καταστρέφει την μηχανή τρόμου η οποία συνθλίβει εδώ και έξι μήνες το λαό της Συρίας. Μιλάμε για 3.000 θύματα τουλάχιστον. Ελπίζω λοιπόν ότι η άσκηση πίεση από το Κοινοβούλιο, τουλάχιστον για μεμονωμένε περιπτώσει, όπω για αυτή τη κυρία Νασέντ, μπορεί να δώσει αποτέλεσμα. Ε, ευνοϊκή έκβαση θέλουμε. Να απελευθερωθεί η κυρία Νασέντ, διότι μιλάμε για μια ψυχαναλήτρια που καταδικάστηκε χωρί λόγο, συνελήφθη χωρί λόγο. Και αυτό προκάλεσε τη διεθνή κατακραυγή. Η γυναίκα αυτή είναι ασθενεί. Η απελευθέρωση τη θα είναι μια νίκη για όλου μα και θα κάνει μια διαφορά θετική αλλαγή για ολόκληρη τη Συρία. Σα ευχαριστούμε. Κυρία Μάισνερ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, εάν καταδικαστεί η κυρία Νασέτ και πραγματικά αυτή είναι μια ένδειξη αυθαιρεσίας, ε, βαρβαρότητας αλλά και παράνοιας του Συριακού κράτους, όπω ήδη ελέγχθη. Γιατί πώς μπορεί να φοβάται ένα κράτος, μια γυναίκα η οποία είναι ηλικιωμένη και άρρωστη και βοηθάει ανθρώπους που έχουν υποστεί ψυχικά τραύματα. Τι είναι εδώ το επικίνδυνο. Τη είπαν ότι έχει αποσταθεροποιητική ε, δράση ως προς το κράτος. Ε, η δικτατορία ε, δίνει εντελώς εσφαλμένα μηνύματα. Η κατάσταση αυτή είναι εντελώς σουρεαλιστική όπως ελέγχθη ήδη εδώ. Ε, όλοι χαιρετήσαμε την Αραβική Άνοιξη και τη διαδικασία εκδημοκρατισμού. Βεβαίω χαιρόμαστε ω Ευρωπαίοι και προσπαθούμε να στηρίξουμε αυτή την Αραβική Άνοιξη. Αλλά θα πρέπει να αγωνιστούμε εάν κάποιοι συλλαμβάνονται χωρί να συντρέχει απολύτω κανένα λόγο γιατί τέτοιο συνιστά κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μάισνερ. Ο κύριος ε, Μικάλσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επιτροπέ, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε εδώ για την περίπτωση ενός και μόνου ανθρώπου, όμως ε, χαίρομαι που στην Ολομέλεια αυτό είναι το σημείο αφετηρίας για να συζητήσουμε όλοι μαζί για την Συρία με αυτή την αφορμή. Το παράδειγμα της κυρίας Νασέντ είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το τι συμβαίνει στη Συρία και τι δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Πάντως, πρέπει να ενώσουμε τις φωνές μας Δεν πρέπει να υπάρχουν διαφωνίε μεταξύ μα. Θα πρέπει όλοι μαζί να καταδικάσουμε τέτοιου είδου συμπεριφορά. Είναι απαράδεκτο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ψώνει το ανάστημά τη. Δεν πρέπει να υπάρχουν πολιτικέ διαιρέσει ω προ το θέμα αυτό σε αυτήν την αίθουσα τη Ολομέλεια. Πρέπει ξεκάθαρα να δηλώσουμε ότι ό,τι συμβαίνει στη Συρία είναι απαράδεκτο. Ευχαριστούμε κύριο Νικολάσικ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι, ε, οι ενέργειες των Συριακών Αρχών κατά των διαδηλωτών και οι πράξεις βία ε, πέφεραν τουλάχιστον 3.000 ε, θύματα, 30.000 θύματα. Οι αρχές 3.000 ε, θύματα, συγγνώμη. Οι ε, αστυνομικέ δυνάμεις ε, πυροβολούν αδιάκριτα κατά των πολιτών. Τέτοιες πράξεις απαιτούν μια καταδίκη εκ μέρου μας. Το ίδιο ισχύει και για αυθαίρετε συλλήψει, συλλήψει χωρίς να υπάρχει απολύτως κανένας λόγος, όπως η σύλληψη της κυρίας Νασέντ οι συλληφθέντες συχνά βασανίζονται από τις αρχές της Συρίας. Γι' αυτό ε, καλούμε τις Συριακές αρχές να τηρήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προβούν άμεσα στην απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων. Κυρία Νταντσίλα, Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποδεχτεί ότι είναι θεμητές οι προσδοκίες των σύρων πολιτών για την μετάβαση προς τη δημοκρατία. Θα πρέπει να σεβαστούμε την επιθυμία τους να ζουν σε συνθήκες ασφάλειας, να ασκούν τα νόμιμα δικαιώματά τους. Η σύλληψη κάποιων πολιτών όπως της κυρίας Νασέντ χωρίς κανέναν ε, προφανή λόγο περιπλέκει την μετάβαση της χώρας προς ένα δημοκρατικό καθεστώς. Και αυτό για τον επιπλέον λόγο ότι οι αρχές της Συρίας δεν φαίνεται να μπορούν να απτύξουν κανένα διάλογο με τον υπόλοιπο δημοκρατικό κόσμο. Πρέπει λοιπόν για να ξεφύγει από την κρίση η Συρία να περάσει σε συζήτηση. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα λόγο μεσολαβητικό ε, με τι αρχέ τη χώρα προκειμένου να αποδεχτούν ότι οφείλουν να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα πρέπει να υπάρξει κοινωνική και οικονομική μεταρρύθμιση. Διότι τέτοιου είδου μονοκινήσει μπορεί να είναι μια μακροπρόθεσμη λύση ώστε να ευνοηθεί το μέλλον τη χώρα και σταθεροποίηση του δημοκρατικού τη πολιτεύματο. Ο δημοκρατικό, η δημοκρατική σταθεροποίηση απαιτεί την άμεση απελευθέρωση τη κυρία Νασέντ. Ευχαριστούμε και τώρα η Επίτροπο μπορεί να απαντήσει. Thank you. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι ξεκάθαρο ότι πολλοί από εσά αναφερθείτε στο γεγονό ότι όλη μα σκέψη είναι στραμμένη προ το Συριακό λαό που συνεχίζει να υποφέρει κάτω από τη βάναυση καταστολή του καθεστώτος του Μπάσαρ Αλασάντ. Επάνω από 3.000 άνθρωποι έχουν φωνευθεί μέχρι στιγμής. Ε, πολλές άλλες χιλιάδες παραμένουν σε κράτηση ε, κάτω από αυθαίρετες συνθήκες σύλληψης και υπόκεινται σε κατάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές οι συλλήψεις και οι κρατήσεις αυτές είναι αδικαιολόγητες και άδικες. Και θα ήθελα να φωτίσω τη συγκεκριμένη περίπτωση της κυρίας Ραφάνα Σέρ, της γνωστής ψυχαναλήτριας της Συρίας, η οποία παραμένει εδώ και έξι εβδομάδες στη φυλακή. Συνελήφθη χωρίς απολύτως κανέναν λόγο παρά την προχωρημένη της ηλικία και την κακή της υγεία. Δεν συνέτρεχε κανένας λόγος για τη σύλληψή της. Είπατε εκπρόσωπος, αντιπρόεδρος, αντέδρασε άμεσα και απίθυνε μια έκκληση για την άμεσα απελευθέρωση της κυρίας ε, Νασέτ μαζί με όλους, με όλους τους άλλους που, έχουν, που κρατούνται παράνομα. Ε, και είναι ξεκάθαρο αγαπητά μέλη θα πρέπει να συνεχίσουμε την πίεση ούτως ώστε να απελευθερωθούν όλοι αυτοί οι αθώοι άνθρωποι συμπεριλαμβάνομενες και της κυρίας ε, Νασέτ. Εμείς έχουμε επιβάλει κάποιες ε, κυρώσεις κατά του καθεστώτος και θα πρέπει να συνεχίσουμε την άσκηση πίεσης για να σταματήσει η βία. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι μέσα των Ηνωμένων Εθνών συνεχίζουμε το έργο μας όσον αφορά την βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία και ένα ειδικό τμήμα του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ένα ψήφισμα για την ε, Συρία με δρυμμή τόνου και αυτό χάρη στη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση για την περίπτωση της κυρίας Ραφάνα Σέτ έχει περατωθεί και μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Θα ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία για πέντε, ε, ψηφίσματα, για πέντε προτάσεις ψηφίσματος για το Θιβέτ, ειδικότερα για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις περιπτώσεις μοναχών.